επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Φαντάλεν, στρατηγική στόχη και συστάσεις πολιτικής για τις θαλάσσιες μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2018. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Φαντάλεν ως εισηγητής για τέσσερα λεπτά. Er Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μπορεί να πει κανείς πολλά για την ευρωπαϊκή πολιτική των μεταφορών αλλά εγώ θα επικεντρωθώ επί δύο βασικών σημείων. Το πρώτο βασικό σημείο είναι η σημασία που έχει ο τομέας. 80% του παγκοσμίου εμπορίου περνάει από τις θαλάσσιες μεταφορές και ο Ευρωπαϊκός τόλο έχει το 41% της παγκόσμιας αυτής αγοράς. Εντό τη Ευρωπαϊκής Αγοράς 40% όλων των αγαθών μεταφέρονται από πλοία. Άρα είναι κρίσιμος οικονομικός τομέα αυτός, κυρία Πρόεδρε, που πρέπει να ανταγωνιστεί σε μια παγκόσμια αγορά. Εάν το καταλάβει κανείς αυτό, τότε το δεύτερο βασικό σημείο συνεπάγεται αυτομάτω. ανταγωνισμός. Ξέρουμε ότι οι χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικού τρόπους για να υποστηρίξουν τους στόλους τους. Αν επιτρέψουμε να γίνει αυτό στην Ευρώπη, θα χρειαστούν μερικά χρόνια μέχρι ότου όλα τα πλοία μα να αλλάξουν σημαία και να αλλάξουν σημαία και να βάλουν σημαία Χονγκ Κόνγκ και Θα μειωθεί έτσι ο στόλος, αλλά και θα επηρεαστεί και όλη η θαλάσσια δραστηριότητα, η απασχόληση, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείε, λιμάνια, ε, εταιρείε επιμελητίας, ε, φορείς εκπαίδευση, εταιρείε που ασχολούνται με την καινοτομία και τη βελτίωση των διαφόρων περιβαλλοντικών πτυχών του τομέα. Όλα αυτά θα υποστούν τεράστιε ζημιές αν μειωθεί ο στόλος μας και φύγουν τα σκάφη μας. Λόγω αυτών των βασικών σημείων, των δύο που ανέφερα, η έκθεσή μου καλεί τα κράτη-μέλη να προωθήσουν τη χρήση τη σημαία τους. Μιλούμε για ευνοϊκά φορολογικά συστήματα με βάση τη χωρητικότητα για τα πλοία σε τόνου και ε, και φορολογικές απαλλαγές για τους πλειοκτήτες και τους ναυτικούς. Οπότε θα μπορούμε έτσι μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσουμε τον τομέα αυτό. Και έχω ένα ερώτημα για τον Επίτροπο σχετικά με αυτό. Πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει κανόνες, προτάσεις για κρατικές ενισχύσεις για, το θαλάσσια, για τα λιμάνια. Αυτή η πρόταση υποτίθεται ότι θα υποβληθεί το φθινόπωρο. Αλλά δεν ξέρω ποιο χρόνο, το φθινόπωρο ποιο έτους. Αυτό που είναι σημαντικό, κατά την άποψή μου, είναι οι κρατικές ενισχύσεις να είναι διαφανείς και να υπάρχει σωστό έλεγχος. Δεν έχει νόημα να υποστηρίζουμε τερματικούς σταθμούς που δεν χρησιμοποιούνται ή λιμάνια που είναι πολύ κοντά γεωγραφικά σε τρίτες χώρες. Ε, θα ήταν ε, σαν να προσπαθούμε κάτι επιματέο. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και κάτι για την παράγραφο 5 του αγγλικού κειμένου που αναφέρεται στις σημαίες ευκαιρίας. Δεν νομίζω ότι η ορολογία αυτή είναι σωστή Υπάρχει μόνο μια καλή λέξη. Πλοία τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές, με χαμηλότερες προδιαγραφές. Δεν θέλουμε σημαίες και πλοία που ε, αγνοούν και παραβιάζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια. Ε, συζητούμε μιλάμε για την ποιότητα της σημαίας και μια φτηνή όπως αποκαλείται σημαία σίγουρα ε, δεν είναι αυτομάτως και σημαία ευκαιρίας. Υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε. Θα πρέπει να γίνει ελκυστικό ο θαλάσσιο τομέα, ο τομέα θαλάσσιων μεταφορών για του νέου. Γυράσκει ο πληθυσμό τη Ευρώπη συνεχώ και χρειαζόμαστε να κάνουμε πολλά περισσότερα για την νεολαία μα, για του νέου μα. Δεν μπορεί να ξεκινήσει κανεί πολύ νωρί. Πρέπει να ξεκινά να του ενημερώνει του νέου για τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών. Και γι' αυτό χαίρομαι, διότι οι πλειοκτήτε ήδη ξεκίνησαν την ενημέρωση των παιδιών στο δημοτικό κιόλα για αυτό που συμβαίνει στον τομέα αυτό όσον αφορά την απασχόληση, την εργασία στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών. Αυτά είναι τα βασικά σημεία και θα ήθελα να επανέλθω σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φαντάλεν. Ο επίτροπο Πίπαλξ έχει το λόγο. Έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη θαυμάσια του έκθεση για αυτό το τόσο πολιτικό θέμα. Η πολιτική θαλασσίων μεταφορών από το 2008 έχει ήδη ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό και στη στρατηγική του 2020 της Κομισιόν και στην πρόταση για μια νέα βίβλο σε σχέση με τα θέματα μεταφορών που επίκειται. Αυτή η πολιτική μεταφορών είναι στο προσκήνιο σημαντικών αλλαγών στην πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναυτιλία είναι μία από, τις, από τα ισχυρά ατού της Ευρώπης και πρέπει εμεί να βασιστούμε σε αυτό το οποίο έχουμε οικοδομήσει στο παρελθόν. Αλλά θα πρέπει να δούμε και το μέλλον. Ο κύριο στόχο μα θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε μια περαιτέρω ενίσχυση στη μακροχρόνια βιωσιμότητα και αποδοτικότητα τη ευρωπαϊκή ναυτιλία. Αυτό σημαίνει αποδοτικά, αποτελεσματικά, ασφαλή και ε, φιλική προ το περιβάλλον μεταφορά στη θάλασσα. Αυτό θα πρέπει να οδηγεί σε θέσεις υψηλού επίπεδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε έρευνα και κοινοτομία στην Ευρώπη. Έχουμε σημαντικούς στόχους και στον τομέα του περιβάλλοντος. Εμείς θέλουμε να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα συνολικές λύσεις όπως η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η στρατηγική μας έχει εκπονηθεί και πριν από την οικονομική κρίση, αλλά παρόλα αυτά που έχουν προκύψει εξακολουθεί να είναι έγκυρη. Θα πρέπει να δώσουμε μια έμφαση και στόχευση στην διατήρηση και στη βελτίωση της διεθνούς τάξης. Δεν θέλουμε να έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό, προστατευτισμό, ε, πλοία τα οποία δεν υπακούν στις προδιαγραφές, ούτε καν πειρατεία. Νομίζουμε λοιπόν ότι ο καλύτερο τρόπο να το επιτύχουμε αυτό είναι μέσω τη συνεργασία στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που είναι ο κύριο εταίρο μα. Εγώ χαιρετίζω τα συμπεράσματα τη Επιτροπή Μετα μεταφορών όπως έχουν παρουσιαστεί και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πολλά από τα θέματα τα οποία γίνεται έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από την Κομισιόν σε πολλές δραστηριότητες για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Όπως αυτή η οποία μειώνει τις διατυπώσεις για τα πλοία και η οποία είναι σημαντική, ε, σημαντική ψηφίδα στην πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άρση των φραγμάτων. Θέλουμε επίσης, των Θέλουμε επίσης να εργαστούμε και στα κοινωνικά θέματα και στην πρωτοβουλία για τα θαλάσσια θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα παρουσιαστούν το 2011 από την Κομισιόν. Θέλω περαιτέρω να αναφερθώ και στις κατευθυντήρες γραμμές για την αυτιλία το 2010. Οι κατευθυντήρες γραμμές του 2004 δεν θα εκπνεύσουν το 2011 ακόμα και η Κομισιόν λέει ότι θα τύχουν αναδεώρησης μέσα στην επταετία τους αυτή. Λόγω της κρίσης και των σοβαρών συνεπειών της για την αυτιλία πρέπει να έχουμε μια επιφυλακτική προσέγγιση. Για τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να αναλάβουμε προετοιμάζουμε μια λεπτομερή στρατηγική την οποία θα διατυπώσουμε και θα ε, δημοσιεύσουμε φέτος το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε του ομιλητέ εξ των πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Κουμουτσάκος πρώτο, για το ΕΛΚ. Δύο λεπτά. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον και με πολύ θετική και είχε σε μένα πολύ θετική ανταπόκριση η ομιλία του κυρίου Επιτρόπου. Γιατί πράγματι η ναυτιλία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός, ζωτικός θα έλεγα τομέας για την ευρωπαϊκή οικονομία και έχει κάθε λόγο η ευρωπαϊκή ένωση να διαφυλάξει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει σε αυτόν τον οικονομικό τομέα αλλά και σαφώς να διατηρήσει υψηλό το επίπεδο των θαλασσίων μεταφορών. αυτή είναι η πρόκληση κύριε πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι πρέπει να κρατήσουμε και τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική και συντονισμένη στρατηγική στις θαλάσσιες μεταφορές. η έκθεση που συζητάμε σήμερα και η οποία υιοθετήθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία στην αρμόδια επιτροπή είναι μια εμπεριστατωμένη έκθεση που κινείται στη σωστή κατεύθυνση και ήδη το κείμενο έτσι όπως έχει χωρίς αλλαγές και ε, μετατροπές νομίζω ότι ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη να έχουμε μια συγκεκριμένη σταθερή γραμμή προς την κατεύθυνση που μόλις είπα. βεβαίως η ευρωπαϊκή ναυτιλία αντιμετωπίζει στις ημέρες μας τρεις μεγάλες προκλήσεις και μια εξωγενή πρόκληση η πρώτη πρόκληση είναι η ανάγκη αύξηση του ανταγωνισμού. είναι γεγονό ότι ο ελεύθερο ανταγωνισμό είναι το οξυγόνο για την ναυτιλία. ταυτόχρονα όμω πολλέ φορέ οι κρατικέ ενισχύσει γίνονται απαραίτητε γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον πολύ συχνά αθέμητο ανταγωνισμό από τρίτε χώρε. συμπέρασμα λοιπόν οι κρατικέ ενισχύσει πρέπει να διατηρηθούν καθώ έχουν συνεισφέρει στη διατήρηση τη ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή ναυτιλία αλλά και τη οικονομία των κρατών μελών δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η ανάγκη ενίσχυση και βελτίωση τη επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο τη ναυτιλίας διότι υπάρχει θεαματική μείωση του αριθμού των νέων που εισέρχονται στο επάγγελμα αλλά και έλλειψη καταρτισμένων ναυτικών. Επομένω, χρειάζεται μια νέα δυναμική πολιτική. Αυτού του δύο τομεί πρέπει οπωσδήποτε να του αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι η έκθεση κινείται στη σωστή κατεύθυνση. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε σοσιαλιστές. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα το γεγονός ότι προβληματιζόμαστε για το μέλλον μιας ναυτιλιακής στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι αυτή η έκθεση θα συμπεριληφθεί και στην έκθεση για το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη και στη Λευκή Βίβλο της Κομισιόν. Η πρόταση της Κομισιόν του 2008 δίνει τους ε, κατευθυντήριους άξονες για το πώς θα έχουμε μια ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο ναυτιλία της Ευρώπης. Και εμείς έχουμε τονίσει ότι αυτό το, αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα οικολογικά πρότυπα και επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και λογικά παγκόσμια κοινωνικά πρότυπα για μια υγεία ναυτιλία. Θέλω να σταθώ σε τρία σημεία μονάχα. Καταρχήν, η ναυτιλία είναι μια φιλική προς το περιβάλλον μορφή μεταφορών. Θα πρέπει λοιπόν και στο μέλλον αυτός ο κλάδος να μπορέσει να είναι ένα από τα όπλα μας για τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Εγώ υποστηρίζω διαρρήδην το να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους πράσινους λιμένες, ακόμα και αν αυτό δεν είναι σημερινό θέμα, αλλά θα θέλουμε να ζητήσουμε από την Κομισιό και το Συμβούλιο να δουν τι μπορεί να επιτευχθεί στο επίπεδο των πρασινών λιμένων. Μου φαίνεται επίσης απαραίτητο να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού κλάδου έναντι άλλων μορφών μεταφορών. Γι' αυτό κατά την άποψή μα είναι σωστό η Κομισιόν να κάνει μια έκθεση αντικτύπου σε σχέση με την περιοχή της ε, Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας σε σχέση με την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο. Εκεί θα πρέπει όμως η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι αυτός ο περιορισμός σε σχέση με τα καύσιμα δεν θα οδηγήσει σε προβλήματα μεταφορών και ανταγωνιστικότητας. Θα ήθελα επίσης να κάνω μια τελευταία παρατήρηση, η οποία είναι πολύ σημαντική για μένα, και αυτό είναι η, η συμπερίληψη των μεγάλων ευρωπαϊκών λιμένων στο σχεδιασμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι οι θαλάσσιοι λιμένες είναι πραγματικά κομβικά σημεία στις μεταφορές και μπορούν να εξασφαλίσουν αυτό το ρόλο τους πλήρως όταν υπάρχει πραγματική διαλειτουργικότητα και όταν ενισχύεται αυτή η διαλειτουργικότητα. Υπάρχει μια μεγάλη σειρά θεμάτων που πρέπει να αναφερθούν εδώ πέρα. Εγώ όμως θα ήθελα να περιοριστώ να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ καλή αυτή η έκθεση και ελπίζω ότι αυτή η τόσο ισχυρή έκθεση δεν θα αλλοιωθεί από τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Η κυρία Σαββισάρα έχει το λόγο. Εάν είναι εδώ, εάν δεν είναι, όχι. Έχουν οι φιλελεύθεροι κάποιον που θα επιθυμούσε να μιλήσει για σας. Η κυρία Πόλσον. Ε, όχι, και Ζήνε Μάισνερ είμαι. Ε, ζήτησα χρονομιλία. Η κυρία Σάβισαρ δεν είναι παρούσα. Έχει υποβάλει γραπτό παρατηρήσει. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω στη θέση τη. Υποτίθεται ότι υπήρχε αγορητής για τους φιλελεύθερους, η κυρία Σαβισάρ. Αν δεν είναι εδώ, θα πάμε στον επόμενο αγορητή και μετά θα δώσω τον λόγο σε εσά. Εντάξει, από ό,τι γνωρίζω, έχω και εγώ χρόνο αγόρευσης ως εισηγήτρια, ως συντονίστρια, συγγνώμη. Η κυρία Σαβισάρ έχει γραπτή παρουσίαση και την υπέβαλε στην Προεδρία την παρέμβασή της. Πάμε στην επόμενη πολιτική ομάδα, στους Πρασίνους. Και μετά εσείς θα έχετε το λόγο κυρία Μάισνερ, εντάξει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέσετ για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα των Ευρωπαίων Πρασίνων υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκθεση και τι συστάσεις του κυρίου Βαντάλεν. Το κείμενο αυτό είναι ισορροπημένο καρπός στενής συνεργασίας που δημιουργήθηκε με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ε, υποστηρίζουμε την λόγω έκθεση διότι θέτει σωστά τα διακυβευόμενα της ε, θαλάσσιας, της πολιτικής θαλασσίων μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλουμε σημαντική αύξηση των θαλασσίων μεταφορών σε διεθνές και ενδοκινοτικό επίπεδο χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον ή τα διάφορα κοινωνικά θέματα. Αυτό το κείμενο εντάσσεται στην ε, λογική που θέλουμε να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, δηλαδή τη λογική βιωσίμου ε, αναπτύξεως. Ανοίγονται θετικοί δρόμοι μέσω του κειμένου, τόσο στις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018, να μπορέσουν να απτυχθούν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η καταπολέμηση των καταχρήσεων της σημαίας ευκαιρίας ή των πλοίων ε, εκτός προδιαγραφών είναι κάτι που θέλουμε να εξεταστεί. Θέλουμε να υπάρξει και προστασία κατά της πειρατείας. Θα πρέπει η πολιτική ε, να εξεταστει θελουμε να υπαρξει και προστασια κατα της πειρατεια θα πρεπει η πολιτικη να ασκηθει σε επίπεδο ενιαίας ευρωπαϊκής Θάλασσα και θα πρέπει να υπάρχουν πολυκομβικέ διασυνδέσεις των λιμένων ε, της Ευρώπης με την Εδοχώρα. Θέλουμε να προστευθούν οι διοικητικοί κανόνε για την είσοδο και έξοδο τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Θα πριν να προωθηθούν τα παγγέλματα, τα σχετικά ανασταλές μεταφορές και η συνεχής κατάρτιση και υποστηρίζουμε και την προτεραιότητα που δίδεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Εν γέννη, ό,τι ακολουθεί την προώθηση των θαλασσίων μεταφορών και να γίνουν ανταγωνιστικό τρόπο μεταφορά, σε συγκρίσει με τι αερομεταφορέ, μεταφορέ, πάντα θα υποστηρίζουμε αυτή την προσέγγιση. Η έκθεση του κυρίου Βαντάλεν ε, λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικές πτυχέ και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές. Μάλλον είναι απάντηση στις προκλήσεις για το περιβάλλον θαλάσσιες μεταφορές. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο τη της αυξήσεως θερμοκρασίας στον πλανήτη. Λυπούμεθα μόνο διότι η τροπολογία που υποβάλαμε με σκοπό οι θαλάσσιες μεταφορές να ενταχθούν στο σύστημα ανταλογών ε, ε, εκπομπών άνθρακος δεν ελήφθη υπόψη, δεν έγινε αποδεκτή από τον εισηγητή ούτε από την Επιτροπή. Κατά την άποψή μας, κανένας οικονομικός τομέας δεν θα πρέπει να εξαιρείται από τον κοινό κανόνα και όπως και αερομεταφορές, όπως και οδικές μεταφορές, έτσι και θαλάσσιες μεταφορές, παρόλο που δεν εκπέμπουν πολύ πολλά αέρια, θα πρέπει να συμβάλλουν όμως την προσπάθεια μειώσεω των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου και θα υποστηρίξουμε στην Ολομέλεια την τροπολογία που υποβάλαμε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριος Χένιν για την ΚΟΕ, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εφημισμό είναι να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια στρατηγική ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα. Αυτό είναι ένα πραγματικά διακυβευόμενο για το μέλλον τη Ένωσή μα σε ό,τι αφορά την τροφιμική ασφάλεια και την ασφάλεια σε ό,τι αφορά τους βασικούς, τα βασικά αγαθά. Για να είναι όμως θετική αυτή η πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει συνολικά τα πάντα, την ε, κατασκευή πλοίων, την επισκευή τους, την κατάρτιση, τη συντήρηση κτλ. Το 2006 η ε, οδηγία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο μας για τους λιμένες και την υποδομή τους είναι ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής στον ναυτιλιακό τομέα. Πρέπει το Κοινοβούλιο ζητά από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να αγωνιστούν κατά των σημαίων ευκαιριών. Αυτό ο αγώνα έχει μόλι ξεκινήσει. Κατά την ουσί... σε επίπεδο ουσία δεν είναι μόνο η καταχρήσει των σημαίων ευκαιρία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά και η ίδια η ύπαρξή του. Γιατί παρά τα καλά και τα ωραία λόγια για την ασφάλεια και τις θέσει εργασία. Αυτά δεν τηρούνται από αυτές τις σημαίες ευκαιρίες. Είναι απαραίτητο να έχουμε σεβασμό στα κριτήρια ποιότητος σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τα κοινωνικά θέματα, να υπάρχει διατήρηση θέσεων εργασίας και καλύτερη κατάρτιση ναυτικών από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η πραγματική στρέβλωση δεν είναι οι κρατικές βοήθειες, αλλά το κοινωνικό dumping το οποίο γίνεται σε μισολογικό επίπεδο και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Ο καλύτερος εγγυητής της ασφάλειας είναι να έχουμε καλοπληρωμένα και καλοεκπαιδευμένα πληρώματα τα οποία να βασίζονται να έχουν καλές συνθήκες εργασίας και καλή κοινωνική κάλυψη. Με ικανοποίηση βλέπω ότι μιλάμε επιτέλους για την διαβίου κατάρτιση των ναυτών, των ναυτικών και βελτίωση των προσόντων τους. Θα πρέπει όμως αυτό να θεωρηθεί ότι είναι ένα δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους στη θάλασσα και κάτι το οποίο πρέπει να χρηματοδοτείται από τους εργοδότες. Εγώ υποστήριζω και τις αιτήσει για τα ναυπηγεία και την ποιότητα του χάλιβος εκεί. Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία στο κείμενο το οποίο μας υπευλήθη, αλλά έχει ακόμα μεγάλες ε, αντιφάσεις γιατί βρίσκεται ακόμα στη βάση του ανταγωνισμού ο οποίος με μεγάλη ελευθερία μπορεί να παρακάμπτεται και ακολουθεί τις ουτοπίες του υπερφιλελεύθερου τρόπου σκέψης. Πώς μπορεί να υπάρξει ας μια έρευνα για να δούμε με ποιο τρόπο οι τεχνολογίες μπορούν να αντικαταστήσουν του εργαζόμενου στη θάλασσα. Πώ θα το υποστηρίξει κανεί αυτό, πώ θα υποστηρίξει κανεί το dumping όταν ζητούμε την ελευθερία κυκλοφορία των εργαζομένων, όταν δεν έχουν ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια δικαιώματα. Πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όταν ορισμένοι δεν διστάζουν να μεταφέρουν προϊόντα τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και για τη φύση και για τους ναυτικούς χωρίς να τα δηλώσουν. Υπάρχουν πολλά ακόμα να πράξουμε, αλλά εμείς πρέπει να αγωνιστούμε για όλα αυτά γιατί είναι απαραίτητο μια ναυτιλιακή πολιτική υψηλού επίπεδου να εξασφαλίσει και το σεβασμό των ανδρών και των γυναικών αυτών που πολλές φορές διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των άλλων. Thank you. Now, Madame Rosbach. Ευχαριστώ η κυρία Ρόσπαχ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φιλόδοξο έγγραφο στρατηγικής, έχω όμως κάποιες παρατηρήσεις. Ε, περισσότερα αγαθά στα μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης, ναι, αλλά τι θα κάνουμε με τη στάθμη του νερού που ήταν ε, πολύ χαμηλή τα τελευταία χρόνια ώστε να μην ε, είναι πλωτή ε, από, από, τα σκάφη που μεταφέρουν τα αγαθά. Και έλεγχος που να βασίζεται στον κίνδυνο. Ναι, αλλά πώς θα βλέπουμε αν γίνεται όταν γίνεται εμπορία ανθρώπων στα πλοία αυτά. πολλά παλιά πλοία τρίτων χωρών μπορούν να υποφεληθούν ε, από τα μέτρα αυτά. Η πειρατεία, γιατί ε, το πρόβλημα αυτό αναφέρεται μόνο όσον αφορά την Αφρική. Ε, στην Ινδονησία το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και αυτό επίσης είναι κάτι που επηρεάζει τις εφοπλιστικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωση. Βρίσκω επίσης λυπηρό το ότι έχουν κλείσει τόσοι μικροί λιμένε. Θα πρέπει να ενισχύσουν ενισχύσουμε την ακτοπλοεία και όχι να την αποδυναμώσουμε. Και μία τελευταία παρατήρηση. Συζητιέται πολύ η σημασία των ναυπηγείων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση όμως σχετικά με την ε, απόσυρση των πλοίων ε, που να γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Η συζήτηση αυτή που γίνεται, ε, διότι στέλνουμε τελικά τα πλοία μας στις Ινδικές ακτές όπου γίνεται ο παροπλισμός των πλοίων με τρόπο καθόλου φιλικό προς το περιβάλλον. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Τα, θέματα των θαλασσίων μεταφορών στην Ευρώπη δεν μπορούν να συζητούνται ξεχωριστά από τα θαλάσσιες μεταφορές στο παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε σε ανταγωνισμό όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών και εμπορευματοκιβωτίων. Λοιπόν, σε αυτό το τομέα θα πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, θα πρέπει να βελτιώσουμε και την κατάρτιση των ναυτικών, ε, να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών, θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε και τις συνθήκες διαβίωσής τους όταν αυτοί είναι στη στεριά. Ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών της Ευρώπης, ξεκινώντας από τον τομέα της ε, ναυπηγικής και εκείνο που χρησιμοποιούν ε, τα σκάφη, ο τομέας υποφέρει από τα ειδικευμένα χέρια οι Ασιάτες, οι Μέση Ανατολή έχουν, ε, παρέχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από ότι οι εταιρείε ευρωπαϊκές. Και σε αυτό το τομέα οι επαγγελματίες των θαλασσίων μεταφορών προτιμούν ε, ναυλωτές του Ντουμπάι, της Κίνας και θέλουν να ταξιδεύουν οι ναυτικοί με άλλη σημαία. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά, ούτως ώστε να υπάρξει μια εναρμόνιση ε, των μέτρων στον τομέα, να, υπάρχει μαθητή, να προβλέπονται μέτρα μαθητή στον τομέα, να βελτιωθεί η παιδεία, η εκπαίδευση ε, στον τομέα των θρασίων μεταφορών. Άλλο θέμα είναι η ασφάλεια που καμιά φορά θέτει σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία των θαλασσίων μεταφορών, των διεθνών θαλασσίων μεταφορών. Ξέρουμε τι συμβαίνει κοντά στο κέρας της Αφρικής. Η Αταλάντη, η επιχείρηση Αταλάντα είναι μια επιτυχία, αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια θα πρέπει οι στατιωτικοί να έχουν ε, σκάφη με πολύ καλύτερες επιδόσεις από αυτά που έχουν τώρα στη διάθεσή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ελκαντράου έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο κύριος Φλέκενστάιν και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή έκθεσή του. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία τονίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν. Καταρχήν η σημασία της ναυτιλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει να κάνει με τον παγκόσμιο ρόλο της Ευρώπης στον εμπορικό επίπεδο και επίσης την δυνατότητα, την ανάγκη να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, αλλά συγχρονώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το αϊφόρο της ναυτιλίας, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπίσουν στον τομέα του περιβάλλοντο. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για όλου. Αυτό σημαίνει ότι οι κρατικέ επιδοτήσει θα πρέπει να ξεπεραστούν. Ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο η απασχόληση και οι συνθήκες εργασίας των ναυτικών θα πρέπει να γίνει και πάλι ελκυστικό αυτό το επάγγελμα για τους νέους. Είναι βέβαια δύσκολο αυτό. Πρέπει όμως να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες, να δώσουμε τις κατάλληλες πληροφορίες στους νέους για τις καριέρες που μπορούν να ακολουθήσουν. Και επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε σημαντικά τις συνθήκες εργασίας στα πλοία να τηρηθούν τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και να υπάρξει πλήρης αστυνόμευση της εφαρμογής της, τους και κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ναυτιλία είναι πράγματι ένας τομέας <clears throat> ο οποίος μπορεί να έχει δυνητικό χαρακτήρα ως αηφόρα μορφή μεταφοράς, αλλά μπορούμε ακόμα να επιφέρουμε πολλές βελτιώσεις, ιδίως με τη συνεργασία στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Επίσης θα γίνει ελκυστικό το ναυτικό επάγγελμα όταν εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στα σκάφη. Πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν σαν πακέτο και εδώ μπορεί να τονίσει κανεί τη σημασία να υποστηριχθεί και η αποστολή Αταλάντα στην Σομαλία. Κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν ως πρώτη ομιλήτρια από την ε, ομάδα Άλτε να ευχαριστήσω τον κύριο Φαντάλεν ε, που έχει δώσει την ψυχή του για το θέμα των, ε, της ναυτιλίας. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του θέματος αυτού. Η ναυτιλιακή οικονομία τα τελευταία χρόνια πριν την κρίση αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο από άλλους τομείς της οικονομίας και οι θαλάσσιες μεταφορές παίζουν σημαντικό ρόλο και είναι σημαντικό το θέμα αυτό για το μέλλον της Ευρώπης. Υπάρχουν και οι προβλέψεις ότι μετά την ε, κρίση θα ξαναναπτυχθεί ο τομέας των μεταφορών ε, και ε, μεγάλη σημασία θα έχει ο τομέας της ναυτιλίας. Το 90% των μεταφορών των αγαθών μας περνάνε από τα λιμάνια και θα πρέπει να θα πρέπει να έχουμε ανθρώπους που να θέλουν να εργαστούν στον τομέα αυτών, οι οποίοι να έχουν ε, ε, καλή εκπαίδευση και η οποία να είναι συντονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι νέοι θα πρέπει να δούνε και ότι υπάρχουν ευκαιρίες στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Και ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να υπάρξει αντικείμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρθηκε και το περιβάλλον. Η εναυτιλία είναι φιλική προ το περιβάλλον, ιδιαίτερα όσον αφορά τι εκπομπέ ε, διοξιδίου του άνθρακα. Μπορεί να βελτιωθεί όσον αφορά ε, το άζωτο και το θείο, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε πάνω στο θέμα αυτό και ο ίδιο ο τομέα και εμεί στην Ευρώπη. Διότι, όπω ήδη υπόθηκε και είναι σημαντικό αυτό, οι θαλάσσιε μεταφορέ σε διεθνές επίπεδο είναι ε, αντικείμενο ανταγωνισμού. Η, η Ευρώπη έχει η ε, ηγετική θέση και θα πρέπει να τη διατηρήσουμε αυτήν. Και θα πρέπει να φροντίσουμε μαζί να αναπτύξουμε περαιτέρω τον τομέα αυτών. Πρόκειται για τομέα του μέλλοντος και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μια καλή στρατηγική. Ευχαριστώ κύριε Μάιστερ. Ο κύριος Ρίκετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είναι πρωταρχή σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να σκηθεί μια πολιτική θαλασσίων μεταφορών που είναι φιλόδοξη και έχει μακροπρόθεσμου στόχου. Και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι ιδιαιτερότητε του τομέα και να απαντά στι προκλήσει που αντιμετωπίζονται. Οι θαλάσσιε μεταφορέ είναι ένα τομέα στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση από πολλέ πλευρέ καταρχάς λόγω του ρόλου που διαδραματίζει στην ανάπτυξη και την απασχόληση, λόγω της διεθνούς διαστάσεώς του, λόγω του χαρακτήρα του του οικολογικού και του βιώσιμου. Υπενθυμίστηκε ότι 80% των εμπορικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο μεταφέρει και οι ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκθεση του κ. Βαντάλεν δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί και καθορίζουν στόχου στρατηγικού και εντοπίζει τους βασικούς τομείς δράσεως για την πολιτική των θαλασσίων μεταφορών της Ενώσεως. Θα ήθελα από την πλευρά μου να επιμείνω επί κάποιων σημείων που υποστηρίξαμε τη συνάδελφό μου την κυρία Βλάστο στην Επιτροπή Μεταφορών για να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των θαλασσίων μεταφορών και κάτι τέτοιο περνά από τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και τις δυνατότητες καριέρας που προσφέρονται στον τομέα χωρίς ο στόχο της ανταγωνιστικότητας να αποσυνδέεται από αυτόν της βιώσιμης ανάπτυξης του θεμητού ανταγωνισμού και της ασφαλείας. Όσον αφορά το περιβάλλον, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προωθεί την εσωτερική του εξωτερικού κόστους και θα πρέπει να υπάρχουν θαλάσσιες ζώνες ελέγχου των εκπομπών. Όσον αφορά την αύξηση των θασίων μεταφορών, χρειάζονται επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό και την αύξηση των υποδομών των λιμένων. Αυτό πρέπει να υποστηριχθεί. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από σήμερα να προωθήσει αυτό το όραμα για την πολιτική στον τομέα αυτό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μέχρι το 2018 η έξοχη έκθεση του κ. Βαντάλεν που υποστηρίχθηκε ευρέω εντό τη επιτροπή. ελπίζω ότι θα υποστηριχθεί εξίσου σε μεγάλο ποσοστό και στην Ολομέλεια και αυτό θα μας δώσει μεγάλη ισχύ στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρίκετ. Την κυρία Τσικάου έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει μεγάλη σημασία η λαυτιλιακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα τομέα όμω ο οποίο αντιμετωπίζει μια μεγάλη, ένα μεγάλο ανταγωνισμό όχι μόνο σε ενδοευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξού και η ανάγκη να υποστηρίξουμε όλες τις πτυχές της ναυτιλιακής πολιτικής και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν πολλά σκάφη τα οποία βρίσκονται σε μαύρη λίστα και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πείσουμε τους εφοπλιστές να καθαρίσουν από τη μαύρη λίστα τα πλοία αυτά και να τα αναβαθμίσουν. Επίσης, Είχαμε πολλά ναυτικά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει σε όλα τα παράκτια κράτη-μέλη κέντρα παρέμβασης, ευρωπαϊκά κέντρα παρέμβαση σε περίπτωση ναυτικών καταστροφών. Κύριε Επίτροπε, εγώ εκμεταλλεύω αυτή τη συζήτηση για να σας επαναλάβω την αίτησή μου η Κομισιόν να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την άμεση πρόσβαση που έχει πιάσει στη Μαύρη Θάλασσα που είναι μια σημαντική στρατηγική σημασία θάλασσα και να υπάρξει μια αντιμετώπιση αντίστοιχη με αυτή άλλων θαλασσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρξουν αιτήσει υποβολής προγραμμάτων για να δημιουργηθούν διάδρομοι στην Μαύρη Θάλασσα. Με τον Ρήνο, τον ε, Μάρνη και τον ε, Δούναβη μπορούμε να έχουμε ε, διαδρομές που να μειώνουν σημαντικά τον δρόμο που πρέπει να διατρέξουν τα πλοία τα ευρωπαϊκά από την Βαλτική στον, ε, στη Μαύρη Θάλασσα. Η θαλάσσια μεταφορά είναι λιγότερη παντική από όλε μορφέ μεταφορών, γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να περιληφθεί και η ναυτιλία μέσα στο σύστημα εμπορία εκπομπών. Επίση, πρέπει να τονίσουμε τι δυσκολίε που έχουν τα ναυπηγεία μέσα στο πλαίσιο τη κρίση, γι' αυτό οι εκπρόσωποι των ε, ναυπηγείων τονίζουν ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται μέσα στην κρίση. Όλο και περισσότερο υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, οι συνθήκες εργασίας και την διακόπτη την ομιλήτρια ο πρόεδρος. Όλα αυτά είναι σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού στόλου και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερη κινητικότητα των ναυτικών, χωρίς κανένα εμπόδιο. Σας παρακαλώ να παραμείνετε στο χρόνο σας. Δεν βλέπω τον κύριο Κέλλιν στην αίθουσα. Θα δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Αγιάλα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον κύριο Βάνδαλο, κύριο Βαντάλε συγγνώμη, για αυτή τη θαυμάσια πρωτοβουλία που δείχνει την ε, θέληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσει στα θέματα της ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που ο κ. Βαντάλεν δέχτηκε πολλέ από τι προτάσει μου. Η έκθεση είναι πολύ σημαντική, υπερλαμβάνει την ανάγκη να υπάρξει αναβάθμιση των σκαφών και των λιμένων και αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων που έχουν αναπηρίε. Επίση, η προσαρμογή στα πρότυπα του Διεθνού ε, Ναυτιλιακού Οργανισμού και εφαρμογή σε όλο τον ναυτιλιακό κλάδο. Επίση, η επαγγελματική κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα του ναυτικού επαγγέλματο για να μην υπάρχει εκμετάλλευση και υποβάθμιση του επαγγέλματο. Επίση, τονίζει να παίξουμε ένα ρόλο ο οποίο είναι ηγετικό <clears throat> για την προστασία από τη ρήπανση, για την χρήση καλύτερων καυσίμων, ιδίω αυτών που είναι πιο φτωχά σε θείο. Παρακαλώ. Νόμιζα ότι μου είχατε κόψει το μικρόφωνο επίσης θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε ευφυά μέτρα μεταφοράς όπως είναι ο Γαλιλαίος και άλλα συστήματα πλοήσεις με δορυφόρο. Είναι απαραίτητο επίσης να αντιμετωπιστεί η πειρατεία και να ενισχύσουμε την δράση Αταλάντα στην περιοχή της Σομαλίας και επίσης να έχουμε καλύτερη ε, σχεδίαση των πλοίων για να εξασφαλίζουν την ασφαλειά τους. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνουν και λιμάνες στα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα και η σύνδεσή τους με τα εσωτερικά λιμάνια και με άλλους κόμβους μεταφορών. Ευχαριστώ. Διαδικασία Καστιάε. Ο κύριος Παπα-Νικολάου πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά φιλόδοξη η στρατηγική που συζητάμε σήμερα και όσον αφορά τις βασικές κατευθύνσεις έχω πλήρως καλυφθεί από την εισήγηση του κυρίου κουμουτσάκου που είναι και ο ε, εισηγητής της δικής μας πολιτικής ομάδος. επιτρέψτε μου όμως να κάνω μια παρατήρηση και ως μέλος της επιτροπής ΛΥΜΠΕ σε σχέση με την πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιας παρακολούθησης με την επωνυμία e maritime. συγκεκριμένα σύμφωνα με το κείμενο τη επιτροπής προβλέπεται η δημιουργία ενό ολοκληρωμένου συστήματο διαχείριση πληροφοριών το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα αναγνώρισης παρακολούθησης εντοπισμού και αναφοράς όλων των πλοίων που βρίσκονται στη θάλασσα και των φορτίων τους. παρόμοιες όμως ηλεκτρονικές δράσεις παρακολούθησης δεν ξέρω αν είναι πιο ανεπτυγμένες ή λιγότερο αναλαμβάνουν και οι δυνάμεις της frontex στο πλαίσιο για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. θέλω λοιπόν να ε, ρωτήσω κατά πόσο αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας αν πρέπει να διευκρινίσει κάτι η επιτροπή στην ανακοίνωσή της αν πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορετικές αρμοδιότητες σε κάθε φορέα ή μήπως πρέπει αυτές οι πληροφορίες να συγκεραστούν ούτως ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και για τις δύο κατευθύνσεις. Ευχαριστώ πολύ. τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα που ανέφερε ο εισηγητής, αλλά δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα είναι η πειρατεία. Οι συστάσεις είναι πολύ καλές, αλλά πολύ γενικόλογες. Ίσως η εμπειρία μας θα έπρεπε να συμβάλλει περισσότερο στους κανόνες για την προστασία που προβλέπει το Διεθνής Οργανισμός ε, ναυτιλία βάσει των εμπειριών από την επιχείρηση Αταλάντα, διότι πιθανότατα θα αυξηθεί η πειρατεία και θα επεκταθεί. Και η Ένωσή μα δεν μπορεί να αποραπλασιάσει τέτοιε επιχειρήσει σε όλο το θαλάσσιο χώρο που χρησιμοποιεί το εμπορικό, εμπορικό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δεύτερον, χρειάζεται πιο λεπτομερή διασύνδεση μεταξύ των εσωτερική ναυσιπλοεία και θαλασσίων μεταφορών, διότι είναι πολύ περίπλοκη η δραστηριότητά μα αυτού του τομεί. Αυτό το δείχνει και η διασύνδεση μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών παραγόντων του, της, ε, του Ευξήνου Πόντου και του Δούναβη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πάσκου. Η κυρία Τικάου σήκωσε τα χέρια της. Μιλήσατε, αλλά αν θέλετε προσθέσετε κάτι, ορίστε. Ναι κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από τον ε, Επίτροπο δύο ερωτήσεις να υποβάλω. Πρώτα απ' όλα, σχετικά, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια έκθεση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του προγράμματος Μάρκο Πόλο. Δεύτερο ερώτημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξει νέα πρόταση νομοθετικού περιεχομένου όσον αφορά το ρόλο των θαλασσίων λιμένων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην όλη οργάνωση την ναυτική σε παγκόσμιο επίπεδο του ναυτιλιακού τομέα και την επιμελητία. Ε, νομίζω ότι έχουμε κι άλλον έναν αγορητή. Ο κ. Κουμουτσάκος έχει το λόγο που μου δίνετε το λόγο τον ξαναζήτησα για ένα μόνο λόγο διότι στην εισήγησή μου την αρχική έκανα μια παράληψη και είναι κάτι που δεν ακούστηκε και από τους άλλους συναδέλφους εδώ. Θα ήθελα εδώ να πω για τον ρόλο της EMSA, της European Maritime Safety Agency. Κάνει ένα σπουδαίο έργο, είχαμε την ευκαιρία με άλλους συναδέλφους να την επισκεφθούμε πρόσφατα, κάνει ένα σπουδαίο έργο, πολύ χρήσιμο για την ανάπτυξη της στρατηγικής των θαλασσίων μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται την υποστήριξή μας και πιστεύω ότι τα στοιχεία και οι τεχνικές δυνατότητες που έχει όχι μόνο βοηθούν την ε, ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές της Ένωση, αλλά μπορούν να βοηθήσουν και σε άλλους τομείς όπως πριν λιγάκι υπόθηκε και κυρίω όσον αφορά παραδείγματο χάρη στοιχεία που μπορεί να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει και η frontex ειλικρινά και κλείνω με αυτό η εμσα κάνει ένα σημαντικό έργο και πρέπει να το γνωρίζουμε και να το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μιλάμε και για τη θαλάσσια στρατηγική της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Thank you. Now, Commissioner, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ήρθε η ώρα σας να απαντήσετε. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που σίγουρα ενισχύει την έξοχη έκθεση του κ. Βαντάλεν και νομίζω ότι είναι πολύ καλογραμμένη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο να συντάξει μια έκθεση γενική, έκθεση για τη στρατηγική, διότι η στρατηγική είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο που έχει μακροπρόθεσμο όραμα και ταυτόχρονα πρέπει να επικεντρώνεται επί βασικών σημείων. Ε, εργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προετοιμάζουμε λεπτομερή οδικό χάρτη για την εφαρμογή των μέτρων, αναμένεται το θέρος να υποβληθεί. Θα ήθελα να απαντήσω σε τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Για τις προσανατολισμούς, για τις κρατικές ενισχύσεις στους λιμένες ήταν μια ερώτηση. Το συζητούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση περί ανταγωνισμού. Έχουμε τον Επίτροπο για Ανταγωνισμό και ό, προσπαθούμε να συνεργαστούμε οι επίτροποι, διάφοροι συναρμόδιοι επίτροποι. Δεν μπορώ να δώσω ε, ε, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δουλεύουμε. Όσον αφορά το Μάρκο Πόλο, το συζητήσαμε το θέμα σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Λοιπόν, η συζήτηση για το Μάρκο Πόλο θα σχετιστεί με αυτά τα δίκτυα. Όσον αφορά τους θαλασσίους λιμένες, δεν έχουμε σε αυτή τη φάση δρομολογήσει κάποια νομοθεσία, δεν έχουμε προετοιμάσει κάποια νομοθεσία. Ξανά ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ αξιότιμα μέλη για τη συζήτηση. Πάρα πολύ βοηθάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συζήτηση. Ήταν πολύ επικοδομητική. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, κύριε Επίτροπε. Και τώρα ο κ. Μαντάλεν, ο έχει το λόγο. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι καλό παράδειγμα καλή συνεργασίας ανάμεσα στι διάφορε πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία βασικά θέματα τα οποία αναφέραν κάποιοι από εσά. Το περιβάλλον είναι ζωτική σημασία. Διότι ο τομέα της ναυτιλίας πρέπει να είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον. Σκέφτομαι για παράδειγμα τα τέλη στα καύσιμα, που έχουν χαμηλό περιβαλλοντικό προφίλ. Σκέφτομαι μήπω θα ήθελε η Κομισιόν να, σκεφτεί την πρόταση αυτή. Και επίσης αναφέρθηκαν οι πράσινοι λιμένες. Νομίζω ότι και αυτό είναι καλή ιδέα. Με άλλα λόγια, ένα πλοίο φιλικό προς το, το περιβάλλον να περνάει πιο γρήγορα από τις διαδικασίες και να πληρώνει χαμηλότερα τέλη. Και αυτό θα ήταν καλή ιδέα. νομίζω ότι είναι θετικό αυτό το κίνητρο, το, ε, αν κάποιος έχει ε, καλό περιβαλλοντικό προφίλ να ε, ανταμείβεται. Νομίζω ότι αυτή είναι εξαιρετική ιδέα και Όσον αφορά την ασφάλεια, ένα από του συναδέλφου το ανέφερε αυτό ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε το τρίτο πακέτο τη ναυτιλία πολύ γρήγορα στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι σημαντικό. Η κυρία Θήκα ανέφερε το μνημόνιο κατανόηση του Παρισιού και έχετε δίκιο ότι αλλάζουν οι επιθεωρήσει, βασίζονται στον κίνδυνο ε, παρά σε ένα σταθερό ποσοστό. Και πάλι λοιπόν ε, ε, ανταμείβεται η καλή συμπεριφορά και θα ήθελα να αναφερθώ στη Σλοβακία που δεν βρίσκεται ακόμα στο λευκό κατάλογο. Παρακαλώ λοιπόν να καταβληθούν πλέον προσπάθειες. Και μιλήσαμε και για τη συντήρηση των πλοίων. Ξέρουμε, την κατασκευή και συντήρηση. Ξέρουμε ότι όσον αφορά την, τα, τα γραφεία ταξινόμησης, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά όσον αφορά το θέμα αυτό, διότι θέλουμε να φροντίσουμε να μην χαθούν θέσεις απασχόλησης. Και τέλος, η αποστολή Αταλάντα. Πρόσφατα το, ο στόλος ε, της Ολλανδία απελευθέρωσε πλοίο από του ε, πειρατέ. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να επιφέρουμε προσθέμενη αξία με την αποστολή αυτή. Τέλο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο και την Επιτροπή στο σύνολό τη και ελπίζω όλε οι συστάσει να ενσωματωθούν στον οδικό χάρτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φαντάλεν. Τελείωσε η συζήτηση για αυτό το σημείο. Η ψηφοφορία θα γίνει σε δύο εβδομάδε. Κατά τη διάρκεια τη ολομέλεια μα στι Βρυξέλλε. Καλωσορίζω την Επιτρόπη κυρία Κρούς και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης.